Κλείνουμε την ημερήσια διάταξη, λέει ο Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε τι εξή ανακοινώσει. Στην 5η 6 Δεκεμβρίου από 9 μέχρι 10 θα έχουμε κοινή συνεδρίαση ΕΚΟΝ και ΕΝΒΗ για την ταξινόμηση βιώσιμη άμα χρηματοδότηση και από 10 έως 12 θα έχουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με ατζέντα, την ψηφοφορία για το MPL και την ακρόαση με τον πρόεδρο των Συνδύ. Στο 3 έχουμε την αναφορά για τις ε, διαθεσμικές διαπραγματεύσεις για το REFIT. Συνέχιση των διαπραγματεύσεων λοιπόν για την, ε, την εξαίρεση από τα ταμεία συνταξής και προκαταρτικές συζητήσεις για θέματα όπως η αρχή της ε, δίκαιης πρόσβασης για τις ε, οντότητες ε, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εκτιμώ το γεγονός ότι αναφέρεται με λεπτό τρόπο ότι δεν έχουμε βρει ακόμα συμφωνία. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το Συμβούλιο να μετακινηθεί. Επόμενο σημείο. Σχέδιο γνωμοδότησης και τον, για την Ο κ. Φρουτζούλικα είναι ο εισηγητής και έχει και το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και Στα ρουμανικά, φροντζουλίκα και φροντζουλίτσα το ίδιο σημαίνουν, αλλά ξέρετε, οι Ρουμάνοι έχουν ως βάση λατινική γλώσσες φροντζουλίκα. Όχι φροντζουλίτσα, δεν είναι σλάβικο το όνομα. Σας ευχαριστώ. Μετά από τόσα χρόνια ήθελα πραγματικά να σας εξηγήσω πώς προφέρετε το όνομά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να με συμπεθάτε. Αγαπητοί συνάδελφοι. να ξεκινήσω τονίζοντας τη σημασία των ε, απαλλαγών σε ό,τι αφορά τις τρεις ε, εποπτικές αρχές ΕΣΜΑ, ΕΟΠΑ και ΕΠΑ. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να εντοπίσουμε ενδεχόμενα προβλήματα και να κάνουμε και προτάσεις για βελτιώσεις. Επιπλέον, θα ήθελα να καλωσορίσω τις συστάσεις του Αλλακτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις οποίες οι συναλλαγές ε, για τους ετήσιους λογαριασμούς, καθώς και η σχετική έλεγχη είναι τακτική. Σε ό,τι αφορά την ΕΠΑ, την ΕΣΜΑ και την ΕΙΟΠΑ, έχουν το καθήκον της ενοποίησης της αγοράς και έχουν και στόχο την προστασία, συστημική σταθερότητα και προστασίας του συστήματος. Θα ήθελα να τονίσω λοιπόν το κεντρικό ρόλο των αρχών για να εξασφαλίσουν ότι θα λειτουργήσει καλύτερα το οικονομικό σύστημα σε ό,τι αφορά και την εθνική υποπτία. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, τα εισοδήματα τα εθνικά θα μειωθούν μετά την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν λύσει για τη χρηματοδότηση γιατί μόνον υπάρχουν επαρκέ πόροι θα μπορούν ε, οι εθνικές αρχές να κάνουν σωστή χρηματοδότηση. Και μετά από την απόφαση της 20 2017 σε ό,τι αφορά την ΕΠΑ, σε ό,τι αφορά τη μετατόπιση στο Παρίσι, την επεκατάσταση στο Παρίσι, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες για το πώς αποφασίστηκε αυτή η μετακόμιση. Αυτά έχει η ζωή. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στις ε, επιπτώσεις που θα έχει αυτό στον προϋπολογισμό. Τονίσω την ανάγκη να υπάρχουν πιο πολλές, ε, πολλά κονδύλια για την καταπολέμηση ναι. του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Να γίνουν και σχετικές ε, έρευνες για εθνικές αρχές. Στο πλαίσιο των, ε, των διαπραγματεύσεων, συμφωνώ ότι θα πρέπει να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος από παράνομες πηγές. Η ΕΠΑ σε σχέση με την ΕΣΜΑ και την ΕΟΠΑ θα πρέπει να βρει τρόπους να ενσηματώσει τους κινδύνους AML και στην εποπτεία και στον έλεγχο. Σε ό,τι αφορά την ΕΣΜΑ, να τονίσω ότι ο, χρημα... ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται 42% άμεσα από τις ε, συνεισφορές των κρατών μελών, 29% από τις ε, τέλη των των ε, οργανισμών και 2% από άλλες πηγές. Πιστεύω ότι αυτές οι ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση μπορούν να απειλήσουν την ανεξαρτησία των οργανισμών. Και αυτό ισχύει και για τον ΕΙΟΠΑ. Ο προπολογισμό είναι 40% από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και 60% με άμεσες συνεισφορές από τα κράτη-μέλη. Και άρα υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για πιο στενή παρακολούθηση σε κάποια κράτη-μέλη για να αντιμετωπιστούν ε, σημεία ευάλωτα και να προστατευτούν οι καταναλωτές από αδίκες, αθέμητες πρακτικές πολύ εθνικών ομίλων. Πολλά είναι τα παραδείγματα που πολλούν, ε, κάνουν πωλήσει ασφαλιστικών προϊόντων σε χώρες της κεντροευρωπαϊκής ε, στην Κεντρική Ευρώπη προϊόντα χαμηλή και τέλος, οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να επιδεικνύουν καλύτερη διαφάνεια, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο, αλλά και προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί σας για να πετύχουμε μια καλή συμφωνία σε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα για την οικονομική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η βάση της έκθεσης των τριών ε, εκθέσεων είναι η εξέταση, η έρευνα του ελεκτικού συνεδρίου. Και θα ήθελα να τονίσω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε ικανοποιημένοι με το ελεκτικό συνεδρίο. Εξ όσων εκτιμώ, αυτές οι εκτιμήσεις και οι αξιολογήσεις του ελεκτικού συνεδρίου είναι πολύ επιφανειακές και διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τα αρνητικά στοιχεία. Ε, θεωρώ ότι είναι τα ίδια. Στον ΙΟΠΑ, για παράδειγμα, θεωρούμε ότι σε ό,τι αφορά τα, ε, συνολικά, τα σημαντικά στοιχεία είναι, λέει, αντικειμενικά. Το ίδιο λέμε για την ΕΣΜΑ. Δηλαδή για τα υπόλοιπα, τα μη σημαντικά, δεν είναι αντικειμενικές οι εκτιμήσει του, Και στην ΕΟΠΑ αναφέρεται επίση. σε όλα τα σημαντικά ζητήματα. Συνολικά υπάρχει αντικειμενικότητα. Αλλά οι πληροφορίε που υποβάλλονται αφήνουν πολλά ζητήματα εκκρεμή, πολλά ερωτηματικά και θα πρέπει να πραγματευτούμε και το περιεχόμενο σε ό,τι αφορά τις ε, συμβατικές, για παράδειγμα, πληρωμές, ε, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, ε, διαγωνισμούς για πρόσληψη προσωπικού που δημοσιεύονται σε ό,τι αφορά τις ε, δημόσιες προμήθειας. Γίνονται παρατηρήσεις από το ελεκτικό συνέδριο, αλλά το συνολικό αποτέλεσμα είναι πενταθετικό. Μα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Πώς να κάνουμε τέτοια, να χορηγήσουμε απαλλαγή. Θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε αυτό από τεχνικής άποψης πιο καλά από ότι το ελεκτικό συνέδριο. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατηρήση. Δεύτερη παρατηρήση τώρα για τις προτάσεις του συναδέλφου Βρουντζουλικά, ο οποίος και στις τρεις ε, οργανώσεις, στους τρεις οργανισμούς αναφέρει τα ίδια στοιχεία, όλα τα ταυτόσημα. Μόνο η ονομασία αλλάζει μόνο σε ό,τι αφορά την εποπτεία των τραπεζών. Υπάρχει ένα έκτο σημείο ότι το 2019 ο οργανισμός θα φύγει από τον Έμενα Βασίλειο και ότι αυτό θα έχει επιπτώσει στο προϋπολογισμό. Έχω σημαντικές αμφιβολίες κατά πόσον αυτό αποτελεί πραγματικά την ουσία του ελέγχου μας. αναφέρει διάφορα για το καθήκον των οργανισμών, έχοντας υπόψη και τον ΑΙΟΠΑ. Κάνει... Πρώτα ψάχνει διάφορες απαγορεύσεις, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις προμήθειες, αν δεν εκτελεί το έργο το οποίο της έχει αναθέσει το νομοθέτημα. Και στο σημείο 4 του συναδέλφου τονίζει ότι και οι τρεις οργανώσεις πέρα από τις υφιστάμενες αρμοδιότητες που έχουν, χρειάζονται επιπλέον αρμοδιότητες για την καταπολέμηση νομιμοποίησης παράνομων εισόδων. Αυτό δεν ήταν, ούτε είναι θμήμα των αρμοδιοτήτων τους και θα καταθέσω ανάλογες τροπολογίες τις επόμενες ημέρες. αυτή η γνωμοδότηση αυτή ουσιαστικά δεν τη χρειαζόμαστε. Τι δεν επαρκεί, τόσο απλή που είναι και αφελής. Ευχαριστώ. Thank you for the... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα του ECR. Καλωσορίζω τον νέο μέλος, τον Ραλφ Πάκετ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Ραλφ Πάκετ είμαι. Διάδοχο του κ. Λούνας που έγινε υπουργό Άμυνας του Βελγίου. Προσβλέπω στην μαζί σας όχι μόνο για αυτά τα τρία θέματα που δεν είναι και τα πιο πολιτικώς ευαίσθητα αλλά πρέπει να διεκπεριωθούν παρά αυτά. Για την εντολή του υποπτικού φορέα και το πλαίσιο ε, είναι ικανοποιητικά όλα αυτά και ο προπολογισμό και το προσωπικό μπορεί να ενισχυθεί η διατύπωση. Εκτιμώ και την αναφορά στην καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Το 2018 είχαμε πολλές σχετικές εξελίξεις και εξακολουθούμε να έχουμε εξελίξεις. Διαβάσαμε επίσης τι έγινε στην Deutsche Bank την περασμένη εβδομάδα και ο εισηγητής τονίζει το ρόλο της EBA ε, που παίζει σημαντικό ρόλο στις αρχές αυτές, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σεπτεμβρίου. Τραπεζική αρχή. Θα εξετάσουμε την κάθε ε, παράγραφο όσον αφορά το EML και το CTF, που δεν είναι η ώρα ούτε ο χρόνος να συζητήσουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εξουσίες για το EML και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Αρχής. Και η διατύπωση για τον Brexit είναι καλή και για τη χρηματοδότηση των εποπτικών φορέων. Και προσβλέπω στην συνεργασία με όλους σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπορεί να είναι πολιτικά ευαίσθητο το θέμα. Ο Βολφ Κλίμς από την Άλτε. Ευχαριστώ και εγώ είμαι τακτικό μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και φυσικά η απαλλαγή στην Επιτροπή αυτή είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο εξετάζουμε πολύ προσεκτικά. Όπως είπε και ο κ. Βέρνερ Λάγκε, θα είμαι σύντομος γιατί αυτό που λείπει θεωρώ είναι το εξής. Τον τελευταίο καιρό, δυστυχώς, έχουμε δει τόσο πολλές απάτες, φόρο αποφυγή, φορολογικά εγκλήματα, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Όλο αυτό τι, τι σημαίνει, ότι δεν έχουμε κάνει όσο θα πρέπει να έχουμε κάνει σε θέματα εποπτείας. Και η παρατήρηση ότι αυτό ουσιαστικά είναι ευθύνη των κρατών μελών, δεν επαρκεί γιατί σκοπός και καθήκον της, ε, των οργανισμών αυτών είναι να εξασφαλίζουν μέσω του συντονισμού ότι θα αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα. Αυτό δεν το βλέπω ούτε στην έκθεση, ούτε το σχολίασε ε, το ελεκτικό συνέδριο και θεωρώ ότι θα πρέπει να το ε, περιλάβουμε αυτό. Επίσης, θα ήθελα και πιο πολλές πληροφορίες σε ό,τι αφορά ε, την κατάσταση της ΕΜΠΑ από το Λονδίνο στο Παρίσι. Τι ακριβώς θα σημαίνει αυτό για το προσωπικό, για τα έξοδα. Αυτά θα ζητηθούν κατά πάσα πιθανότητα του χρόνου. Σε ό,τι αφορά την ΕΣΜΑ τώρα, το επόμενο έτος θα σημαίνει τις πιο πολλές αλλαγές. Σε ό,τι αφορά την ΑΙΟΠΑ, το είπε ο Βερνελάγκα, πρέπει να αξιολογήσουν πιο πολλά εσωτερικά μοντέλα που χρησιμοποιούν οι εταιρείε. Και αυτό είναι ένα τομέα όπου ενδεχομένω θα πρέπει να δείξουμε πιο πολύ επιφυλακτικότητα. Συνολικά, η συνεργασία μεταξύ των τριών υπηρεσιών και των ε, εθνικών αρμόδιων αρχών δεν είναι στο σημείο που θα έπρεπε να είναι. Και στον έλεγχο των ε, υπηρεσιών ένα μεγάλο πακέτο το οποίο ελπίζουμε να το συμπληρώσουμε, να το ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος της θετίας, θα πρέπει να φροντίσουμε αυτή ακριβώς η συνεργασία να προσαρμοστεί και να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση των οργανισμών αυτών χωρίς ωστόσο να αποθαρρύνουμε τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Thank you. I don't see Ευχαριστώ, δεν βλέπω τον Sven Giegold. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους πρασίνους θα μιλήσει εκ μέρους του. Θα μιλήσει κάποιος για το Σβέν Γκίγκολτ ή πάμε στην επόμενη ομάδα. Ουδέμια απάντηση. Άρα η απάντηση ομαδα μια απαντηση όχι. Από τους άλλες, άλλες ομάδες δεν βλέπω κάποιον. Πάμε στο Catch the Eye. Η Περβάνος Περέζ έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Αυτή η έκθεση Αυτές οι εκθέσεις για την απαλλαγή είναι σημαντικές και χαίρομαι τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού εμβαθύνει στο έργο της. Θα πρέπει να προσέξουμε ούτω ώστε αυτές οι εκθέσεις περί απαλλαγών να μην γίνουν εκθέσεις όπου καλύπτουν τα πάντα. Εισάγονται πτυχές που θέλουμε να αναφερθούν. Το λέω αυτός αυτό προφανώς αναφερόμενοι σε δύο στοιχεία που αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Πώς αυτοί οι οργανισμοί, η ταπεζική αρχή των αρχών, των αγορών και της ασφάλειας, των ασφαλίσεων, θα παρεύουν για το ξέπλυμα του χρήματος και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι θέματα υποσυζήτηση. Και αυτό γίνεται στα πλαίσια της εκθέσεως που προσπαθώ μαζί με τον Μακάρας να περάσουμε, να ψηφιστεί και δεν θα πρέπει όμως να προδικάσουμε αυτό το θέμα προς στα πλαίσια της απαλλαγής. Αν το κάνουμε αυτό, βλάπτουμε την δελεχή εξέταση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά αυτή την πρόταση, και ο πρόεδρος της Επιτροπής Τάξη 2 θα πρέπει να εκκλείσετε από τα συμπεράσματά μας. Υπήρξε συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών. Αυτή όμως δεν αρκεί για να εξασφαλίσει επαρκή εποπτεία του φαινομένου του ξεπλήματος χρήματος. Το ίδιο όσον αφορά την εσωτερική προσέγγιση, το εσωτερικό μοντέλο. Θα το συζητήσουμε στα πλαίσια Τη αναθεωρήσεως των ΕΣΑ, κατά πόσο η ΕΟΠΑ θα έχει περισσότερο ρόλο, ενισχυμένο ρόλο, είναι θέμα αρμοδιοτήτων. Δεν είναι θέμα ορθής διαχείρισης από την ΑΕΟΠΑ του προπολογισμού της. Προτείνω να είμαστε σοβαροί και να βαθύνουμε στα θέματα του προπολογισμού και το πώς χρησιμοποιούνται τα χρήματα από τις αρχές αυτές και να μην αναμειγνύουμε όμως τα άλλα στοιχεία, διότι έγινε αυτό θα υπονομεύσουμε α, τις συζητήσεις επί της ουσίας στις άλλες εκθέσεις της Επιτροπής. Thank you. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Επομένως, κύριε Φρουντσουλίκα και συμπαθάτε με για το λάθος το όνομά σας. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ πρόεδρε γιατί... Κύριε πρόεδρος ξέρετε όσο, όσο γερνάμε κάνουμε το ίδιο και τα ίδια λάθη. Όχι, δεν είναι λάθος, λέει ο κύριος Φουντσούλικα. Ε, απλώ σα το είπα γιατί θεώρησα ότι ω Ιταλό θα με νιώσετε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να σα πω την αλήθεια. Εκπλήσωμαι. Γιατί ο κύριο Λάγκ ήταν πολύ επικριτικό. Ξέρετε, Τα τελευταία χρόνια ποτέ, ποτέ για τις τρεις απαλλαγέ των ειδικών οργάνων δεν ε, είπαμε τέτοια πράγματα. Γιατί τα τελευταία χρόνια η ίδια δομή υπήρχε σε όλες τις απαλλαγέ, Πρόκειται για απαλλαγέ. Και ξέρετε τι λένε οι σύμβουλοι μας. 1500 γράμματα λένε. συμπεριλαμβανομένου και των καινών διαστημάτων. Γιατί μιλάμε για τα θέματα τα οποία αποτελούν κοινό υλικό για αυτά τα τρία θεσμικά όργανα. Και ε, αν, αν την αντιμετώπιση του τρομοκρατίας, τη συνεργασία, το ξέπλυμα των χρημάτων, και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τέλος πάντων, περιμένω τροπολογίες, περιμένω τροποποίησεις, περιμένω νέες ιδέες, προτάσεις. Πέστε τα όμως, καταλαβαίνω τις επικρίσεις σας, αλλά πέστε και κάτι για την ουσία του πράγματος, τα πραγματικά ζητήματα. Τίποτα δεν άκουσα. Ήταν γενικόλογες επικρίσεις. Είπατε τι δεν λέω, ε, πέστε τι, τι θα πρέπει, πού θα πρέπει να πω περισσότερα. Τελευταία δεκαετία ήταν μία από τα ίδια όλες οι απαλλαγές. Εγώ προσπάθησα να διαφοροποιηθώ. Ε, ε όπα, έμπα, έσμα, για, για όλα τα νέα ταμεία. Για την υπηρεσία που θα πρεπει να πω περισσοτερο τελευταια δεκαετια ηταν μια απο τα ιδια ολες οι απαλλαγες εγω προσπαθησα να διαφοροποιηθω ε οπα εμπα εσμα για ολα τα νεα ταμεια για την υπηρεσια που θα εχει εδρα στο Παρίσι. Πέστε μου κάτι για τα πραγματικά θέματα. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Οπότε έχουμε το εξή χρονοδιάγραμμα. Τροπολογίες 6 12 συζήτηση 10 πρώτου και στην ε, Οικονομική Επιτροπή 4 Δευτέρου η ψηφοφορία. Πάμε τώρα στις ψηφοφορίες. Για να δω, έχω τη λίστα ψηφοφορίας. My group.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 Για να δω τώρα τα χαρτιά μου. Έχετε όμως το λόγο. Πρόεδρε, εκ μέρους των σοσιαλιστών να αναβάλουμε την ψηφοφορία όσον αφορά την ψηφοφορία για το benchmark. Γιατί ακόμα δεν έχουμε διαμορφώσει τις θέσεις μας. Δεν μπορούμε να πάμε σε ψηφοφορία σήμερα για τα benchmarks. Ευχαριστώ. Βλέπω συμφωνή και το ΕΛΚ. Άρα αναβάλλεται αυτή η έκθεση. Για να αρχίσουμε την ψηφοφορία. Πρώτα πρώτα δοκιμή. Ψηφίζουν δοκιμαστικά. bodies. Πέρα ψηφοφορίας. Σας ευχαριστώ. Okay, so we start uh, amendment 6. Ξεκινούμε με την τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Έξι. Για το έξι. Πέρασε. Εγκρίνεται 17-15. Συμβαστική α. Υπέρ κατά εγκρίνεται. Β. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Γ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20. Προφορική τροπολία του εισηγητή ή της εισηγήτριας εγκρίνεται F. Υπέρ κατά εγκρίνεται τροπολογία 26. Υπέρ κατά εγκρίνεται 27. Υπέρ κατά εγκρίνεται 28. Υπέρ κατά εγκρίνεται 29 υπέρ κατά εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 32 υπέρ κατά αποχές, ε, έλεγχος για το 32. Πέρασε. 19-18 εγκρίνεται. 35 συμβατή υπέρ κατά εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά έλεγχος για το 2 ψηφίζουμε Πέρασε. 17-15 εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Εποχή. Τόσο με διαψηφορία αν θέλει να κάνουμε έλεγχο. Αν όχι πάμε στο 37. Συγγνώμη, καταπίπτει. Πάμε στο 38. Διορθώνει ο πρόεδρος. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Έλεγχος για το 41. Ψηφίζουμε. Απορρίπτεται 17-18, 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 43 υπέρ κατά έλεγχος για το 43 ψηφίζουμε. Πέρας εγκρίνεται 20-17. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά έλεγχος για το 44. Πέρας. Εγκρίνεται. 20-15. Το 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας. 32 με 5 αποχές. Ψηφίζουμε για την απόφαση που αφορά τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. η κυρία Τελάνκια Αλτσέσπα δεν έχω την ε, ψήφο, οπότε προσθέστε το, όπως δήλωσε. Όσον αφορά την ε, επίστευση για τον τριμερή διάλογο, ψηφίζουμε. Η νομιστική ψηφοφορία συν η ψήφος κ. Ντελάγκη. Πέρας. 34 συν μία ψήφος. Έχουμε την ειδική ψηφοφορία. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Τώρα πρώτα θα ψηφίσουμε τον κανονισμό. διασυνοριακή κατανομή των συλλογικών πόρων επενδύσεων. Εγκρίνεται. Για να δω που είναι οι τροπολογίες. Τροπολογία 180 υπέρ κατά Α, είναι αυτή η διαβόητη. Αυτή είναι Μάρκος. Υπέρ, κατά. Αποχές, απορρίπτονται. Κοιτάξτε, κάτι διαδικαστικό. Κάναμε την ψηφοφορία. Χωρίς μικρόφωνο, ο δεν ακούει τι λέει στη συνέχεια. Δικαστικό επαναλαμβάνει για να αποφύγουμε τις προστριβές. Δεχτήκαμε, δεχτήκαμε το αίτημα για την ψηφορία, αλλά σας ξεκαθαρίζω ότι οι τροπολογίες του εξή δεν θα είναι παραδεκτές αν δεν αφορούν το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Γιατί αν αρχίσουμε να τροποποιούμε άλλον κανονισμό, δεν, δεν, μας αφορά αυτό τώρα, εκτός από τα σημεία που υπάρχει μια ευρεία συνένεση των ομάδων. Αλλά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε επί άλλων εκθέσεων. Να μην το συζητήσουμε, γιατί το αποφασίζουμε αυτό με ψηφοφορία. Ωραία. Καλά να σας δώσω το λόγο, αν θέλετε. Αλλά αυτό έχω να σας πω στον τι θα κάνω στο μέλλον. Εάν δεν υπάρχει ευρεία συνένεση των πολιτικών ομάδων, τότε θα κηρύσσεται απαράδεκτη η νέα τροπολογία, η οποία δεν θα αφορά ε, τον, τον εν λόγω κανονισμό με την ε, ε, αποφασιστή σαν νομική βάση κλπ. Μπράιν, εγώ θέλω απλώς να πω μπράβο που μας τα είπες αυτά, πρόεδρε, που τα αποφάσεις, γιατί ε, τώρα διαμορφώνουμε την πραγματικότητα όπως δεν γίνει ποτέ στο παρελθόν σε αυτό το επίπεδο. Γιατί μέχρι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο δεν γινόντουσαν τέτοια πράγματα. Οπότε μπράβο, μπράβο, μας δίνει ευκαιρία να ψηφίσουμε. Και έτσι τώρα υπάρχει ασφάλεια και υπάρχει βεβαιότητα για την κατάσταση πραγματική. Την επόμενη φορά που θα φέρει πρόταση η Κομισιόν, τότε, ε, τότε μπορεί να καλύψουν όλα τα σχετικά και να μην ε, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την κερκόπορτα του δεύτερου πυλώνα που από νομοθετική πλευρά είναι φάουλ. Καλά λέει ο πρόεδρο. να συνεχίσουμε την ε, ψηφορία. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουν την ε, από τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ε, ψηφορία συν Α, όχι, κύριε τώρα έχει την, την κάρτα, συγγνώμη. Πέρα ψηφοφορίας. 34 υπέρ, 0 κατά, 5 αποχές. Ψηφίζουμε τώρα την απόφαση να ξεκινήσουμε τις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Ονομαστική Πέρα Πέρας ψηφοφορίας. 33-1 5 εποχές. Έχουμε την ε, προβλεπόμενη ψηφία για τον τριμερή διάλογο. Μπράβο στον εισηγητή. Θα δοθεί η εντολή για την ευρωπαϊκή ψηφορία. Τώρα έχουμε πρώτη, πρώτη συμβαστική. Ε, D. Σελίδα 11. D. Υπερκατά αποχής εγκρίνεται. Θα ψήσουμε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως... Ε, Τροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία, Πέρας. 34-3. Δύο εποχές. Απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων, ονομαστική ψηφοφορία. Ερασοφορίες. 33, 4 είναι δύο εποχές. Συγχαρητήρια, εισηγητά. Είπαμε ότι αναβάλουμε το νούμερο 10 για τα benchmarks. Και τώρα πάμε στην έκθεση TANG. Κοινό σύστημα για τον φόρο ψηφιακών υπηρεσιών όσον αφορά τα εισοδήματα από την παροχή συγκεκριμένων ψηφιακών υπηρεσιών 31-32. Ονομαστική ψηφοφορία. Να έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, υπέρ. Μάλλον άρχεται η ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. τέσσερις ψήφοι εναντίον, 4 υπέρ, συμβαστική α, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 140 υπέρ κατά έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 έλεγχος. Vote Πέρας. 20 ψήφοι κατά, 19 υπέρ, απορρίπτεται. 25 υπέρ, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία. Vote Πέρας. Εγκρίνεται 24-15, 156 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται 20-19 συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 23-16 166-167 υπέρ κατά Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Η διαφορά είναι μικρή, οπότε ας ελέγξουμε. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 20-19. Καλά που ελέγξαμε. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά έλεγχος. υπερας Εγκρίνεται 20-19. 170 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 171 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 173 και 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά φιλελεύθερη. Έλεγχος, έλεγχος. Να σηκώνετε τα χέρια παρακαλώ. Πέρας εγκρίνεται. 21-15, 41 υπέρ κατά Έλεγχος για τη 41 άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, εγκρίνεται. Ένα υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την ένα. Πέρας. Εγκρίνεται. 20-19. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται 71 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτωται 72 υπέρ, κατά αποχές εγκρίν, απορρίπτωται, συμβαστική L υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική M υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 78 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτωται 79 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική N υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά έλεγχος για την 90 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 20-19. Συμβαστική P υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 103 υπέρ κα... έλεγχος για την 103. Άρχεται. Πέρας. 1623 Τροπολογία 104 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 105 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 107 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 14 υπέρ, κατά έλεγχος για 14, ερχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 20-19, 15 υπέρ, κατά έλεγχος για την 15 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας 20-19, 108 υπέρ, κατά έλεγχος για την 108 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας 20-19 εγκρίνεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που τροποποιήθηκε με νομοστική ψηφοφορία. Πάρχεται. Πέρας. 33 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Πρέπει να ψηφίσουμε κάποια παράγραφο του νομοθετικού ψηφίσματος προτείνω όλους μαζί να προτείνουμε. Από 33 μέχρι 39 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτονται. Το νομοθετικό ψήφισμα θεωρείται συγκεκριμένο ως ετροποποίηθη. Πάμε στην έκθεση Ροζάτη. πρέπει να διαβάσει τον τίτλο. Σημαντική ψηφιακή παρουσία. Ο τίτλος τροπολογία 15 ονομαστική ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. 36 ψήφοι κατά μία υπέρ απορρίπτεται. καταγράφεται ότι ψηφίσατε υπέρ της τροπολογίας σας. 62 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 65 υπέρ κατά, υπέρ κατά έλεγχος για την 65. Πέρας 20-19 εγκρίνεται 67, 68, 69 υπέρ κατά έλεγχος για αυτές, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20-19 εγκρίνονται, 79 περ κατά έλεγχος. Πέρας. 20, 19 εγκρίνονται. 80 υπέρ. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 19, 19 απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 83, 84 και 9 υπέρ, κατά έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20-17. Εγκρίνονται. 85 και 86 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνονται. 87 υπέρ, κατά Έλεγχος για την 87. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 20-19. 88. Καταπίπτει. 89. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 89. Πέρας. Ισοψηφία 19-19 απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 92 έλεγχος. Για την 91 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται 21-18. 92 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται 93 υπέρ, κατά έλεγχος για την 93, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται 20-19, 95 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 96 και 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 12 υπέρ, κατά έλεγχος για τη 12, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 21-18, τροπολογία 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γιώτα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20-19, 116 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται 16-19. Συμβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά έλεγχος άρχεται πέρας απορρίπτεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική σ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 20-19. 37. τα 39. Υπέρ. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 20, 19, 41 τώρα. Υπέρ. Έλεγχος. Για την 41 παρακαλώ έλεγχουμε. Πέρασε. Απορρίπτεται 19-20. D, παρακαλώ, συμβαστική D. Δέλτα υπέρ, κατά αποχέ συγκρινεται Συμβαστική E, ε. Όχι, πρέπει να ψηφίσουμε ξεχωριστά. Την 109 πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ δεν είναι στον κατάλογο των σοσιαλιστών. Για την 16 νέα ευαζολή, 109 τροπολογία. Υποθέτω ότι υπορψηφίζουμε. τη των αναλογιών. Δεν είμαι και σίγουρος όμως. Η 109. Δεν ξέρω γιατί άλλαξε η σειρά. Όπως και να έχει, ψηφίζουμε την 109 τώρα. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 ψήφι, κατά 18 υπέρ. 46. 46. Και εδώ θα κάνουμε έλεγχο για την 46. Ψηφίζουμε παρακαλώ πάλι τροπολογία Εύα Είναι ακόμα ανοιχτή η ψηφοφορία για τη 46. Πέρας. Απορρίπτεται. 19 κατά 17 υπέρ. Και τώρα πάμε στη συμβαστική ε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη 46. Όχι, την ψηφίσαμε. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 και 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε παρακαλώ την 61. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται 19 υπέρ 20 Καταψηφίζουμε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αποστροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση έναρξη. Και πέρασε. 36 υπέρ, μία ψήφος κατά, δύο αποχές. Και τώρα να ψηφίσουμε μπλοκ στην 16, 17 και 18. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το ψήφισμα λοιπόν εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα περνάμε στην ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού. Συμβιβαστική α. Υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Και πέρασε. Απορρέπτεται σε ψηφία. Υπέρ. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά έλεγχος ψηφίζουμε παρακαλώ Vote is closed. Uh, reject. Πέρας απορρίπτεται. 34. Συμβαστική έψιλον. Ε. Υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. F. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. Ισοψηφία απορρίπτεται. Η G υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. H ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική G. Ε, H υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 69 παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Είσαστε κατά, μάλιστα. Πέρασε. Εγκρίνεται 23 υπέρ 15 κατά. Αποσύρεται. 98 99 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Κάπα υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Λ υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Μ, εμ υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά. Ψηφίζουμε, ελέγχουμε παρακαλώ την 107. Πέρας. Εγκρίνεται. 23 υπέρ, 15 κατά, νη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική W υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 117 υπέρ, κατά, έλεγχος. Πέρασε. Εγκρίνεται. 23 υπέρ 15 κατά. 108. Μετά θα μπει. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για την 120. Πέρασε. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για 128 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ για 129 έλεγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Σεμιβαστική πι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 136. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 136 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. σεμιβαστική Q. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά Έλεγχο για την 147 παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. 150 υπέρ. Κατά. Έλεγχο. για την 150. Πέρασε. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για την 152 εδώ χρειάζεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 153 υπέρ. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται. 154 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 159 υπέρ κατά. Το ΕΡΚ είναι κατά. Απορρίπτεται. 160 υπέρ κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. 161 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρασε. Εγκρίνεται. 162 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 162 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 163 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για την 163 παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 165. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Πέρας. Εγκρίνεται 166 υπέρ. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική αίσθηση υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 173 υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τάφ. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική γιου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 190. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Έλεγχο για την 185. Πέρας. Εγκρίνεται. 187 υπέρ. αποχέσεις, Απορρίπτεται. 192 υπέρ. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 197 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 198 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. 199 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Σι, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική δι, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 201, 211 υπέρ, κατά έλεγχος παρακαλώ. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 212 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 214 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική D α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 218 υπέρ κατά έλεγχος για την 218 παρακαλώ ελέγχουμε έναρξη και πέρας απορρίπτεται 220 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 221 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Ατυλογική σκέψη 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά έλεγχος παρακαλώ. Πέρας, εγκρινέται. Και την τρία ψηφίζουμε, μάλιστα. Τροπολογία τρία υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέρας. Απορριβέται. τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές εγκρινέται. 4 και 5 αιτιολογικές σκέψεις μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και να προτείνουμε όλες τις λογικέ σκέψεις από την 6 μέχρι και την 10 μαζί. Αν συμφωνείτε υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ. Έλεγχο παρακαλώ την τροπολογία 7. Πέρας. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10. Έλεγχος παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται λογική σκέψη. Τροπολογία 12 μάλλον υπέρ. Κατά. Έλεγχο παρακαλώ. Πέρα. Απορρίπτεται. 13. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 16. Υπέρ. Κατά. Άλτε. 16 εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Έλεγχος την 17. Πέρασε. Εγκρίνεται. Είναι τα παραγράφος 1 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε εγκρίνεται. Είναι τα παράγραφο 2, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα παράγραφο 3, υπέρ κατά αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε. Ναι, ναι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Είναι τα 4. 4.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 Έλεγχος, παρακαλώ, για την άγκρη 6. Πέρας Εγκρίνανται 28-7 υπέρτα. Εγκρίνεται 28 7 υπέρ κατά. Ελέγχουμε. Ψηφίζουμε. Πέρας. 28 εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, Παραγραφός 10 εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το 12 καλύπτεται όχι ψηφίζουμε 12 υπέρ κατά έλεγχος για το 12 ψηφίζουμε Vote is closed. Πέρασε. Απορρίπτεται. 20-18. Ε, επόμενη άκρη 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά έλεγχος για την 15 γεωργίες πέρας εγκρίνεται 18 άκρη 16 υπέρ κατά αποχές ε, ε, ελέγχουμε το την τροπολογία 16 της άκρης πέρας της ψηφοφορίας. Η ισοπαλία 19-19 απορρίπτεται. 17 της Επιτροπής Γεωργίας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Άγκρι 18 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 ε, ναι, υπέρ, κατά, έλεγχος. Ψηφίζουμε. Πέρασε. Εγκρίνεται. 19-18. Ψηφίζουμε το κείμενο όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική ψηφορία. Ονομαστική, ονομαστική. Υπέρ. Πέρασε ο φοριας 32 32-2 με μία αποχή. Εγκρίνεται το κείμενο. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Η επόμενη συνάντησή μας θα είναι στις 6 Δεκεμβρίου. Έχουμε τότε ψηφοφορίες. Πώς? Όχι, όχι, όχι, αν δεν έρθει να ψηφίσετε δεν θα έρθει ο Άγιος Βασίλης με τα δώρα. Παρακαλώ, ελάτε για την ψηφοφορία. Πέρας της συνεδριάσεως, λοιπόν. Mm. I'm really concerned because